Συνόδων Ολομέλεια ε, για την κοινοβουλευτική έτο 2019. Αυτά θα δημοσιευτούν στον τόπο τη Ολομέλεια και ε, προθεσμία για, τις, ε, για την υποβολή τροπολογιών ω τι 7 σήμερα. Θα ψηφιστούν όλα αυτά 18 Απριλίου το μεσημέρι στι 12. Οι ημερομηνίε είναι οι εξή. 14 έως 17 Ιανουαρίου, 30 έως 31 Ιανουαρίου, 11 ε, ως 14 Φεβρουαρίου, 11 ως 14 Μαρτίου, 25 ως 28 Μαρτίου, 3 και 4 Απριλίου, 15 και 18 Απριλίου, 1η και 4 Ιουλίου, 15 ως 18 Ιουλίου, 16 ως 19 Σεπτεμβρίου, 9 και 10 Οκτωβρίου, 21 και 24 Οκτωβρίου, 13 και 14 Νοεμβρίου, 25 έως 28 Νοεμβρίου 16 έως 19 Δεκεμβρίου 2018 όλα αυτά. 19 συγγνώμη. Διάφορες επιτροπές